Κυρίε και κύριοι, σα ανακοινώνω πω η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στι 20 Σεπτεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4, εξέτασε την εντολή του κυρίου Σέρζιο Γκουτιέρε και αποφάσισε να επιβεβαιώσει την εντολή αυτή από τις 20 Ιουλίου. Υπάρχουν παρατηρήσεις. κάποιο κατά. Όχι, άρα η εντολή αυτή επιβεβαιώνεται οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζήτησε να αναλάβει ο κ.